good I can start meeting again and give you the... Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Καταρχήν να σας αναφέρω τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών. Πρώτον, όσον αφορά οι συγητές και συντάκτες, οι συντονιστές συμφώνησαν όσον αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας να μην αναλάβει δράση. Ε, νούμερο 2. Η πολιετής χρηματοδότηση της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Θαλασσιών Μεταφορών πάλι καμία δράση. Θα ζητήσει όμως να ληφθεί υπόψη η έκθεση αυτή, η υπόψη όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις ε, για την εναρμόνιση των ε, ε, διατάξεων για τα οχήματα και για τον θόρυβο, πάλι καμία δράση. Υπάρχει μια έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Οικονομικών για το μέλλον του ΦΠΑ. Ε, ανακοινώνω ότι η ΕΚΟΝ εκπονεί έκθεση με βάση την πράσινη βίβλο της Κομισιόν που θίγει μεταξύ άλλων ερωτήματα που σχετίζονται με την φορολόγηση των μεταφορών επιβατών. Μέχρι τις 22 Ιουνίου λοιπόν έχουν ερωτηθεί οι συντονιστές αν συμφωνούν ή όχι με την εκπόνηση γνωμοδότησης ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ θα είναι στις 19 Σεπτεμβρίου. Ζητήσαμε λοιπόν από τους συντονιστές να σκεφτούν αν θέλουν να εκπονήσουμε γνωμοδότηση για το θέμα αυτό και να μας ενημερώσουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Όσον αφορά ε, τις ε, μελέτες ε, για το 2011 έχουν συμφωνήσει οι συντονιστές για μια σειρά μελετών για τα επόμενα θέματα. Αξιολόγηση της επιβολής του νόμου και των ελέγχων στην κοινωνική νομοθεσία, τις επιπτώσεις περαιτέρω ε, ελέγχων ε, για τις εκπομπές θείου. Και ε, εδώ θα προσθεθεί και το θέμα των αζωτικών ενώσεων. Επίσης, όσον αφορά το, τον ταχυδρομικό τομέα πακέτων και την αναθεώρηση των διεθνών συμφωνιών. Οι συντονιστές επίσης ε, αποφάσισαν αν υπάρχουν ε, ακόμα πόροι μετά από τις μελέτες αυτές, τότε ε, θα ενημερωθεί και η έκθεση για την Eurovelo. Επίσης έχει... Θα αφήσουμε μια άλλη μελέτη για τις μεταφορές ε, λόγω της ε, οδηγίας ε, για την Ευρωβινιέτα. Όσον αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, έχω ενημερώσει τους συντονιστές σχετικά με τις επιλογές που έχουν να ζητήσουν από την Κομισιόν να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Ζητήσαμε από τους συντονιστές να το γνωρίζουν αυτό και τους καλέσαμε να εξετάσουν εντός των ομάδων τους ε, την δυνατότητα αυτή. Όσον αφορά την επιτροπολογία, θύχθηκαν τρία θέματα. Τα υγρά ε, στις χειραποσκευές ε, επιβατών αεροπλάνων. Αυτό είναι ένα σχέδιο πρότασης της Κομισιόν, καθότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις, ε, ζητήσαμε αντιρρήσεις μέχρι τι 16 Ιουνίου, δεν λάβαμε σχετικές αντιρρήσεις ε, και ε, είναι επίγουσα διαδικασία με έλεγχο. Όσον αφορά τις άδειες των πιλότων, τα τα μέτρα αυτά θα ληφθούν ε, τον Ιούλιο. Οι συντονιστές αποφάσισαν ότι θα πρέπει ένας από τους ηγητές επιτροπολογίας να οριστεί ε, εισηγητής ε, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 εάν προταθεί αντίρρηση στην πρόταση της Κομισιόν και στηριχθεί από την πλειοψηφία. Αλλά επειδή αυτή τη ε, στιγμή δεν έχουμε λάβει την πρόταση αυτή, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα υπάρχει αντίρρηση ή όχι. Όσον αφορά την ε, συνάντηση εμπειρογνώμων ITS, ενημερώθηκαν ε, οι συντονιστές σχετικά με την ε, συνάντηση αυτή των εμπειρογνωμόνων, η οποία ακολουθήθηκε από συνάντηση στο γραφείο της κυρίας Γένσεν. Στα διάφορα. Ε, συμφωνίες Ασφαλείας Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, Καναδά αποφασίστηκε να εξεταστεί το... και Βραζιλίας αποφασίστηκε να εξεταστεί το κείμενο της Κομισιόν σχετικά με την ασφάλεια των αερομεταφορών. Συμφωνήθηκε ότι η διαδικασία από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με τροποποίηση των συμφωνιών αυτών δεν θέτει προηγούμενο για μελλοντικέ συμφωνίε. Ε, ζητήθηκε από την ε, ομάδα ECR συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ε, να εκπονήσει δική της έκθεση σχετικά με τις αερομεταφορές. Οι συντονιστές αποφάσισαν να περιμένουν το αεροπορικό πακέτο του φθινοπόρου εξετάζοντας εναλλακτικέ λύσεις όπως θα ήταν προφορική ερώτηση ή κάτι άλλο συζητήθηκε από τον ε, συντονιστή της ομάδα των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ε, να το συζητήσει με την ομάδα του και να απαντήσει. Σύμβαση των Αθηνών. Θα συζητηθεί τον Ιούλιο. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους συντονιστές σύμφωνα με την, σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου να χωρίσει την, ε, το πακέτο αυτό σε δύο κομμάτια με διαφορετική νομική βάση, το άρθρο 10 και 11. Ε, το θέμα αυτό θα είναι αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ενώ τα υπόλοιπα κομμάτια θα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Μεταφορών. Στην ε, συνάντηση 11, 12, στη συνεδρίαση 11, 12 Ιουλίου θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Σημείωσαν οι συντονιστές ε, σχετικά με το, τις προτάσεις ημερολογίου ε, για τα έτη 2012 και 2013. Ο πρόεδρος υπέδειξε την ανομαλία ότι τον Ιούλιο του 2012 ε, η Ολομέλη θα πραγματοποιηθεί Τρίτη με Παρασκευή ε, και όχι ε, Δευτέρα με Πέμπτη, τον Απρίλιο λόγω, της, λόγω του Ορθόδοξου Πάσχα. Επίσης, λένε το οι σημειώσιμο ότι μετά από έντονη συζήτηση, το οποίο μάλλον δεν αποτελεί καθόλου υπερβολή, το αντίθετο, μετά από μια πολύ έντονη συζήτηση, οι συντονιστές αποφάσισαν να αναβάλουν την ψηφοφορία στην Επιτροπή μέχρι τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου ώστε να ε, επιτραπεί στις ομάδες να εξετάσουν τις 700 τροπολογίες που υπάρχουν και τους ε, σχετικούς συμβιβασμούς ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο βαθμό συνένεση εντό τη επιτροπή. Η ψηφοφορία αυτή λοιπόν θα πραγματοποιηθεί νομίζω 10-11 Οκτωβρίου όσον αφορά ε, τις ε, αερομεταφορές ε, και την ασφάλεια, ζήτησα από τους συντονιστές και από τα μέλη να προσεγγίσουν τους επικεφαλείς των ομάδων τους για να φροντίσουν να εμφανίζεται η έκθεση αυτή στο, στην ε, Ολομέλεια του Ιουλίου. Ξέρουμε ότι ο Αντιπρόεδρος Κάλλας ε, της Επιτροπής θα βρίσκεται στην Ολομέλεια αυτή και η Επιτροπή μας έχει ζητήσει ε, σχετική δήλωση για τα υγρά στις χειραποσκευές και ελπίζουμε αυτή η δήλωση να αποτελέσει μέρος της συζήτησης για την έκθεση Grandes. Και τέλος, οι αποστολές του 2012. Είχαμε μία προσωρινή ε, συμφωνία σχετικά με τις, ε, με τις αποστολές που είχαν προταθεί ε, στο Αμβούργο της κυρίας Μάισνερ από την Άλντι και μία στην Κρήτη του κυρίου Δανέλη από τους σοσιαλιστές και περιμένουμε τώρα μία τρίτη από το ΕΛΚ. Αυτά, μας, ε, αυτά είναι από τους συντονιστές. Υπάρχουν ε, ερωτήσεις σχετικές. Εάν όχι, θεωρώ ότι ε, εγκρίθηκαν αυτά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φιντάντσο, έχετε ένα διαδικαστικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη δήλωση από πλευρά τη Ιταλική Αντιπροσωπεία του ΕΛΚ. Σε λίγα λεπτά θα συγκεντρωθούμε για να ψηφίσουμε μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βραζιλία για την ασφάλεια στην αεροπλοεία. Μετά από πρόσφατε αποφάσει τη Βραζιλία για την υπεώθηση του Τσέζαρη Μπατίστη με την μη έκδοση και μάλιστα μάλιστα την απελευθέρωση αυτού του ατόμου, εγώ και ο συνάδελφος Καντσάν δεν θέλουμε να ψηφίσουμε για αυτή την ε, έκθεση. Βέβαια, σέβομαι την ε, δουλειά της, της και των σχεδόν εισηγητών, τους οποίου εκτιμάμε, αλλά θεωρούμε πως σε αυτή τη φάση το να εγκρίνουμε με μία ψήφο, μία συμφωνία με μια χώρα που τάχθηκε κατά στην ουσία μιας χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ήταν σκόπιμο. Δεν έδωσε απάντηση μάλιστα σε δύο αιτήματα του Ευρωκοινοβουλίου που ζητούσαν την έκδοση του Τσέζαρη Μπατίστη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Φιντάντσε. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ. Το πρώτο είναι να έχετε μαζί τις κάρτες ψηφοφορίας και να τις βάλετε στην σχισμή. Και τώρα φυσικά θα κάνουμε τον ε, συνηθισμένο έλεγχο. Ε, το έλεγχο πάντα προσπαθεί να ψηφίσει με έναν παραπάνω. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία, κάνουμε έναν έλεγχο. Έχετε τις καρτούλες σας. Have you got an assistant who can go and run and find your card? Λοιπόν, άντε, τριχάτε να βρείτε τις κάρτες σας όσοι δεν τις έχετε. Okay. Vote is closed. Ωραία, λοιπόν. Ε, τέλος της δοκιμής. I look to Mrs. Everybody legal, Mrs. Very good. Πολύ ωραία. Όλοι ψηφίσατε σωστά λοιπόν. Τώρα... Κάποιος που δεν έχει την κάρτα του θα ψηφίζει με διανάταση στις ε, χειρός ε, ο κύριος Σασόλ. Εντάξει, μέχρι να βρει την κάρτα σας θα κάνουμε αυτό. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Πρώτη έκθεση του κυρία Τικάου για τη συμφωνία με τη Βραζιλία. Μία ψηφοφορία είναι μόνο. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. It's on κάρτα, με την κάρτα γιατί είναι τελική ψηφοφορία. Μια και έξω. Ε, με την κάρτα, το μηχάνημα, ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. And it's 34 υπέρ μαζί με τον κύριο Σασόλη και ένας κατά. Για να σκεφτώ ποιος είναι αυτός ο ένας και μια αποχή μάλιστα. Δύο κατά, δύο. And no abstentions, that's the... Και καμιά αποχή. Ωραία λοιπόν εγκρίνεται. Μπράβο κύριε Τικάου. Okay tourism report. Where's my... Mr. Fidanza's report. Μάλιστα, πάμε στην έκθεση του κυρίου Φιντάνζα. Για να κάτσει εδώ ο γραμματέας δίπλα να, να, μου... να με καθοδηγεί, να μην κάνουμε λάθος ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφοφορία για την έκθεση ίδιες πρωτοβουλίας για την Ευρώπη ως πρώτη τουριστική προορισμός του κόσμου, μια, ένα νέο πολιτικό πλαίσιο για τον τουρισμό στην Ευρώπη και ο Σφιντάντζα είναι πρώτη τροπολογία, Τικάου, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Δανέλης. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στις παραγράφους τώρα συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρόπολογία 29 μετά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37. Παράγραφος 4. Κυρία Τικάου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38. Μπρέπολ Σφιντάντσα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 δεγκράντες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 γράντες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 με την ε, προφορική τροπολογία που έχετε εδώ από τους πράσινους. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 159 Μαρινέσκου. Το πρώτο ένα έχει καταπέσει, το δεύτερο κομμάτι. Θεωρεί ότι και δικαιώματα σε προστασία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93. για λασέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Α, συγγνώμη, 98 πρώτα. Φιντάντζα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην συμβιβαστική, 9, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115. Μπακ. Ποιο είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 είναι η επόμενη. Αγιάλα Σέντερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. <laughs> Α, βλέπω ότι κουραρχίζουν και κουράζονται ήδη τα μπράτσα σας, συνάδελφοι. Μην ανησυχείτε, 30 σελίδιτες ακόμα έχουμε, δεν τίποτα. Τροπολογία 124. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 122 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 10 και 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Ε, η 147 ψηφίσαμε να το ελέγξουμε, αλλά νόμιζα ότι ήταν ξεκάθαρο. Εν περιπτώσει, ξεκινάμε την ψηφοφορία για το 147. Ε, άντε, λίγο να ξεκουραστούν τα χέρια σας. Ε, ψηφίζουμε στην 147, αρχίζει η ψηφοφορία, τέλος της ψηφοφορίας. Ορίστε. Απορρίφθηκε. Σαφώς. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την 161 παρακαλώ ως προσθήκη. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 172 με προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. δεν έχει καταπέσει. Πάμε στην 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα η λέξη οικολογικός τουρισμός υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται και δεύτερο τμήμα με την τοπική βιοπικιλότητα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1.88.188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 194 μόνο τρεις σηκώσατε τα χεράκια σας ε, λοιπόν ψηφίζουμε για την 194 ψηφίσατε όλοι τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 192 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 199 είναι μια χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα λέει ιδιαίτερα στα, στα νέα κρατημέλη να δίνω όλο το κείμενο χωρίς αυτά τα λόγια. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, βάζουμε το δεύτερο τμήμα στη ψηφοφορία τώρα. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Διακόσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «212. Πρώτο τμήμα, το γεγονός ότι οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρώπη θα δώσουν ε, χώρο, θα, θα δώσουν μέλλον στο και τα λοιπά. Υπέρ που κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα είναι η διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.13 Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, 214 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 215 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 217 υπέρ. Απεσύρθη 216, όλα θέλετε να τα μαθαίνετε. 217 υπέρ, κατά αποχές, 218 είπε κατά αποχές, εγκρίνεται. 219 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 22 Those in favor. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ερχόμαστε στη συμβαστική 27. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 238. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική που 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 249 πέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική υπάρχει 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική 25 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 260 με προφορική τροπολογία την οποία βλέπετε Ψήφι Π Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Α, η τροπολογία 5, ψήφι Π Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 6 που δεν καλύπτεται από το 5, το υπόλοιπο δηλαδή, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 10, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τριολογική σκέψη ε αποσύρεται και αντίστοιχε τροπολογίε. Πάμε στη 19. Ψήφι πε. Τροπολογίε 19. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 20 πε. Κατά αποχέ. Α το ελέγξουμε καλύτερα. Και την 20 ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Has everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Α, τώρα έχουμε γνωμοδοτήσεις. Μάλιστα, πάμε στην παράγραφο 6 της νομοδότης Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς ε, που έχει καταπέσει το προηγούμενο. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 6 της ΣΥΜΚΟ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πού πάμε τώρα. Στην αιτιολογική σκέψη ε πάντα τη ΣΥΜΚΟ στην επόμενη σελίδα Έτσι το βρήκατε όλοι ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε Διάφορα έχουν καταπέσει εδώ λόγω συμβιβασμού. Πάμε κατευθείαν στην Περιφερειακή Επιτροπή τώρα στην παράγραφο 3. Δεν ξέρω. Στη δική σα ε, λίστα από ψηφοφορίες που είναι, στο δικό μου κατάλογο είναι σελίδα 19. Παράγραφος 3. Πού είναι το ΙΤΡΕ 5, γιατί δεν το είδα. Α, το βρήκα. Παράγραφος 5 τη Επιτροπή Βιομηχανία, Ήτρε, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη σελίδα 19 και την παράγραφο 3 της Περιφερειακής Επιτροπής, εντάξει, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Yeah. Then, uh, also falls. Right. Because we adopted amendment 12. Yeah, so it's now paragraph 7. Ε, παράγραφος 7 λοιπόν της περιφερειακής πάντα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 23 πάντα στην περιφερειακή είμαστε ψήφι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Γεωργία, παράγραφος 4. Ψήφι Π. Τι έχετε? Όχι, έχει καταπέσει. Γιατί εγκρίθηκε ο συμβιβασμό 24. Εντάξει, ε, ε, πάμε λοιπόν στην παράγραφο 4 της Επιτροπής Γεωργίας. Ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. Για να σας δω τώρα με την Επιτροπή Γεωργίας τώρα. Επόμενη, 13. Πάντα στην Επιτροπή Γεωργίας, ψήφι πέ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία, αποκαταστάθηκε η αρμονία μας στη σχέση. 18 ε, υπέρ, ε, κατά, εγκρίνεται. Πολιτισμός. Ε, παράγραφος 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Παράγραφος της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, 26 της Επιτροπής Πολιτισμού, παράγραφος πάντα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. As everybody voted, voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 35 in υπέρ, συν όλοι 36, 5 κατά χωρίς αποχές εγκρίνεται συγχαρτήρια κύριε Φιντάντζα. Okay, now then we'll change of... Λοιπόν, αλλάζουμε έγγραφα και ξαναγυρνάμε σελίδα 1 τα καλά νέα είναι ότι είναι η τελευταία ψηφοφορία. Α, προσέξτε συνάδελφοι, αυτό μπορεί να γίνει λίγο περίπλοκο, γιατί στην απέναντι σοφία μας δεν έχουμε μόνο συμβαστικές ε, τροπολογίες, αλλά και ε, ψηφοφορίες κατά τμήματα στις συμβαστικές, που αυτό εμένα με ξεπερνάει, αλλά εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε. Πάμε να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Έτσι τι αποφασιστική. Και είναι και έκθεση ιδέας πρωτοβουλία για την οδική ασφάλεια του κυρίου Κόχ. Έτοιμοι. Πάμε. Παράγραφος 2, τροπολογία 14, ψήφι Π. Κατά, άποχες, εγκρίνεται. Η συμβαστική α, ψήφι Π. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. Στην τροπολογία 23 που είναι προσθήκη με προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. υπέ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Του συγητή. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Και 30 ταυτίζονται. υπέ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. υπέ κατά αποχές εγκρίνεται 32 προσθήκη Π. κατά αποχές εγκρίνεται 34 του κυρίου Βαντάλη ψήφι Π. κατά αποχές απορρίπτεται ορίστε 33 φαγιών προσθήκη Π. κατά αποχές εγκρίνεται η 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 36 παρακαλώ αρχίζει το ηλεκτρονική ψηφοφορία ψήφισατε όλοι πέρας τότε 37 με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 ως προσθήκη ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 προσθήκη με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 41 Υπέ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέξουμε. Είναι της κυρίας Γένσεν. 41 αρχίζει ψηφοφορία τώρα. Και αν ψηφίσετε όλοι, τελειώνει. Μ, απορρίπτεται. Άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε τη 42. Ψήφι πέρα κατά αποχές και αυτό θέλει έλεγχο. Νομίζω ότι είναι το ίδιο αποτέλεσμα, Δεν πάει πάση περιπτώσει ψηφίζουμε τη 42. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, Πέρασα. Το ίδιο. Απορρίπτεται. 44. Ψήφι πέ Κατά. Αποχές. Το ίδιο αποτέλεσμα απορρίπτεται. 45. Υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 μπαχ υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να το ελέγξουμε σας παρακαλώ. Για την 55 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Να απορρίπτεται. 56 ως προσθήκη υπέρ της κυρίας αναλόγα κατά απόχες απορρίπτεται. Συμβιβαστική σύ, υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 61 is next. υπέρ. Ε, ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Προσθήκη είναι αυτή. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Those against. Κατά. Α, θέλετε να την ελέγξουμε τη κυρία Γκρισπέκ. Η τροπολογία 63 αρχίζει τώρα ηλεκτρονική παρήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τότε. Απορρίπτεται. 64. Ως προσθήκη ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική δε. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 ως τα επόμενη στις παραγράφου 19 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 του κυρίου Βαντάλεν ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, επειδή εγκρίθηκε 74, θα πρέπει να ψηφίσουμε, λέει, εδώ την προφορική του κυρίου Μπάξ 77, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 προσθήκη ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Και αυτή η προσθήκη είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 80 καταπίπτει νομίζω λόγω της 82 όπως και 81. Πάμε στα 83. Ψήφι Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την 83 αρχίζει ηλεκτρονική υποληθεύση. Και αν ψηφίσατε όλοι, πέρα. Απορρίπτεται. Η 86. Ψηφί Those against, abstentions adopted. 90. Η 90. Υπέρ. Κατά. 90. Κατά είμαστε. Αποχές απορρίπτεται. Η 88. Υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 89. Υπέρ κατά άποχες. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ τον 89, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Υποπτεύομαι ότι θα είναι 19 υπέρ 22 κατά, αλλά δεν ξέρει κανείς ποτέ τι γίνεται. Πέρας τώρα της ψηφοφορίας. Α, λάθος. Εγκρίθηκε. Η συμβαστική ε. Εδώ είναι ψηφοφορία κατά τμήματα. Είναι σε δύο τμήματα ο συμβιβασμό ε. Το πρώτο είναι όλο το κείμενο εκτό από τη λέξη υποχρεωτικό στην πρώτη γραμμή, obligatory. Θυμάστε για την οφθαλμολογική εξέταση, για τον έλεγχο τη όραση. Σε περίπτωση που δεν καταλάβετε είναι θέμα οπτικό. Είπε κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα είναι μαζί με τη λέξη υποχρεωτική. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 94 είναι η επόμενη. Ε, παράγραφος 21α, ναι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 96 πε κατά άποχες εγκρίνεται 97 σε δύο τμήματα συν προφορική τροπολογία λοιπόν τμήμα πρώτο καλή και τα λοιπά και τα λοιπά κατά της κοπόσεως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα που βλέπετε εδώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η προφορική τώρα τροπολογία που θα μπει 29α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 98 η σημαντικότερη όλων ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Εγώ θέλετε, ναι, καλά. Germany's not going to give you a check, Όχι. 105 του κυρίου Βαντάλεν, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίψετε. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 είναι προσθήκη ψηφίπε κατά αποχές. Αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε σας παρακαλώ. Να ψηφίσουμε για την 101. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αψηφίσατε ολοι όλοι πέρα. απορρίπτεται. 103 ως προσθήκη ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 104 επίσης προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 είναι η επόμενη. Της κυρίας Τσικάου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές Απόση... Ε, ε, ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. 112 είναι προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 τα ίδια Είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 έχει αποσυρθεί. 115 προσθήκη ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 116 με την προφορική τροπολογία. Ψηφίπε. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 117 ψηφίπε. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 118 της κυρίας Ράνερ, την οποία έχει αναλάβει ο κύριος Μπαχ. γιατί βλέπετε, δεν ξέρω τι λέει για τους κανονισμούς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 που ζητά επάλυψη υπέρ κατά άποχες. Αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. 122 αρχίζει η Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 21 κατά απορρίπτεται. 123 those in 123 υπέρ. Κατά αποχές. Να την ελέγξουμε και αυτήν. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 123. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 19 ε, υπέρ 23 κατά. Συμβιβαστική τροπολογία F. Μπις υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 129. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 έχει αποσυρθεί. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 του κυρίου ε, χωρίς τη ψηφοφορία. Πρώτον, το σύνολο του κειμένου, εκτός από τη φράση above a pre-agreed speed limit, πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο ταχύτητας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 137 της κυρίας Ζέλερ. Πάλι χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος, εκτός από τα ποδήλατα με την ε, προφορική ε, τροπολογία, τα ε, ποδήλατα με βοηθητικούς κινητήρες που είναι πιο γρήγορα από 25 χιλιόμετρα την ώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος καταπίπτει επειδή το πρώτο δεν εγκρίθηκε. Ε, συμβαστική τροπολογία H, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 143 είναι η επόμενη που αφορά την ε, παράγραφο 25 της κυρίας Τικάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 140 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 προσθήκη. Υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 154, 155 καταπίπτει, 156 είναι επόμενη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 προσθήκη ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την 159 αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω, κύριε Κούν. Ε, μια χαρά τα καταφέρατε χωρίς τον κύριε Γκρός. Μπορείτε παρακαλώ να αφαιρέσετε την ψήφο ενός από τους αλληλεπληρωτές σας. Έγινε αυτό βλέπω. Ε, πολύ καλά. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 19 υπέρ, 22 κατά. Ε, η επόμενη 163 ως προσθήκη υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 και το δεύτερο μέρος ε, μαζί με την Επιτροπή και. Το πρώτο μέρος λοιπόν χωρίς τις λέξεις αυτές υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος λοιπόν... Ναι, πρέπει να ψηφίσουμε και το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 178, παράγραφος 28α, νέο. 178 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100, αναελέγξουμε την 179, αρχή της ψηφοφορίας για την 179. Το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω. As everybody voted, the vote is closed. Ψηφίσατε όλοι η λήξη της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία I, Ι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε κατευθείαν στη συμβαστική τροπολογία J. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 195 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 196 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 207, 207 είναι η επόμενη. Παράγραφος 34α νέο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε αυτήν, διότι νομίζω ότι εγκρίνεται 207 αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 22 κατά απορρίπτεται. 206, those in favor. 206 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία K. και Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. M. Συμβιβαστική τροπολογία M, όπως Μιχάλης είπε. Όχι. Συγγνώμη, η L. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην μη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική τροπολογία N, νη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ...219 είναι η επόμενη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται ούτως ή άλλως, καταπίπτει, καταπίπτει, που είμαστε τώρα. Στη συμβαστική τροπολογία O, όμικρον. Θέλετε να ελέγξουμε την 223. Ωραία, ελέγχουμε την 223. Την τροπολογία του κυρίου Βαντάλεν. Αρχή της ψηφοφορίας. Has everybody voted? The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Be clear, don't we really compromise? Oh. Συμβαστική τροπολογία O, όμικρον. Where was the result? Well, 13 in favor, 27 against. 13 υπέρ, 27 κατά. Ήταν το αποτέλεσμα. Είμαστε ικανοποιημένοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στη συμβαστική τροπολογία. Ο, όμικρον, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη είναι η 228, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 229. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 231. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε μία προφορική τροπολογία του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.33 και 2.34 είναι όμοιες, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 2.32 είναι προσθήκη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία π. Αυτή είναι πολύπλοκη. Ωραία. Συμβαστική τροπολογία π. είναι σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος λέει ότι καλεί τα κράτη-μέλη μαζί με το σημείο 1 μέχρι εκεί που λέει Vehicle Occupants Compulsory. Το δεύτερο μέρος καλεί τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνει τους ποδηλάτες ιδιαίτερα τη νύχτα να φορούν ε, <clears throat> ε, κράνη. Και το τρίτο μέρος ε, καλεί τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνει τους ε, ποδηλάτες, ιδιαίτερα τη νύχτα ε, έξω από αστικές περιοχές, να φορούν γυλαίκα φωσφορίζοντα για να φαίνονται καλύτερα. Πρώτο μέρος λοιπόν της τροπολογίας αυτής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το τρίτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 240 next as an addition. 240 ως προσθήκη, υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.37 ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την 2.37 αρχή της ψηφοφορίας. Τη Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.45 είναι η επόμενη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Q υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.48 ως προσθήκη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.50 ως προσθήκη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.51, χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος είναι το Road Maintenance Workers. Το δεύτερο μέρος αφαιρεί το κομμάτι The Use of Road Safety Barriers with Smooth Surfaces και το τρίτο μέρος είναι το, το υπόλοιπο. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μέρος το υπόλοιπο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία R. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την 259 της κυρίας Κρίσπεκ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 19 υπέρ, 22 κατά. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 260 υπέρ. Ε, αρχή της ψηφοφορίας, συγγνώμη. Ψηφίσατε όλοι, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 20 υπέρ, 21 ψηφί κατά.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 12 και 13 είναι όμοιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τελική ψήφος αρχή της ψηφοφορίας. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια Κυρικό. Συνάδελφοι, έτσι ολοκληρώνουμε τις ψηφοφορίες. Να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και που τα καταφέραμε. Ευχαριστώ και το προσωπικό, διότι είναι πολύ πλοκος αυτός ο κατάλογος της ψηφοφορία. Τους ευχαριστώ λοιπόν. Το επόμενο θέμα μας είναι για την ΕΜΣΑ. Τι ώρα το είχαμε προγραμματίσει αυτό. Η Κομισιόν είναι παρούσα για το θέμα της ΕΜΣΑ. Να προτείνω 10 λεπτά διάλειμμα και να επανέλθουμε στις 10.30. Στο μεταξύ θα προσπαθούμε να βρούμε την Κομισιόν. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Λάχρη θα επανέλθει. Δέκα λεπτά διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε στις μισή αν βρούμε την Επιτροπή. Okay, colleagues, next Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επόμενο θέμα στη μέση διάταξη είναι ο κανονισμός για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φλέκενστάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί από την περασμένη φορά που τα είπαμε δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτά που σας είχα πει τώρα έχουν ε, τότε έχουν γίνει σήμερα τροπολογίες. Μέχρι τώρα συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ θετικέ εμπειρίε που έχουμε αποκομίσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ΕΜΣΑ, και συμφωνώ με που λένε ότι θα πρέπει να προσέχουμε και το κόστος όταν είμαστε στριμωγμένοι οικονομικά αλλά είναι πραγματικές οι συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν στον ε, ΕΜΣΑ και αυτό θα γίνει μόνο εφόσον και όταν ε, το Συμβούλιο μοιράζει όχι μόνο αρμοδιότητες στον οργανισμό, αλλά καταλαβαίνουν και οι υπουργοί όταν γεννούν σπίτια τους ότι αυτό έχει επίδραση και στην εργασία τους εντός των χωρών τους. Έχουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες, μια σειρά τροπολογιών. Η σημαντικότερη και πιο επίμαχη απέναντι στο Συμβούλιο είναι η υπόθεση της πρόληψης και της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρήπανσης και να μην αφορά μόνο ε, πλοία και πετρελοκυλίδες και ρήπανση, αλλά και εξέδρες εξόριξης και ενδεχομένω και άλλα πράγματα όπως ε, ανεμογεννήτριες, ολικά πάρκα κλπ. Όταν μιλάμε για ε, αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, ε, ποιος θα ελέγχει όλα αυτά και ποιος φροντίζει να διατηρούνται καθαρές οι θάλασσες. Έχουμε λοιπόν και πολλές τρεπολογίες που αφορούν την παροχή συμβουλών στα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ενιαία Ευρωπαϊκή Θάλασσα και την κατάργηση της γραφειοκρατίας, το σχέδιο Blue Belt ε, που το ίδιο το Συμβούλιο αποφάσισε πέρσι το Δεκέμβριο στην Ελληνική Προεδρία. Και το θέμα είναι πόσο είναι συμβατό το ε, δίκτυο πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοείας με το SafeSeaNet, τι γίνεται με την πιστοποίηση των αναγνωρισμένων ε, υπηρεσιών και οργανισμών και νομίζω ότι ο οργανισμός αυτός ασφάλειας της θάλασσας μπορεί να βοηθήσει για την κατάρτιση ε, των ναυτικών, διότι με βάση των εμπειριών τους στις σχολές ε, ναυτικών και εκτός της Ένωσης μπορούν να βοηθήσουν και με τις βεύτιες πρακτικές. Κάτι άλλο που δεχτήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να το συζητήσω εγώ, ε, ήταν να διαβρεθεί αυτό το θέμα και σε γείτονε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη βοήθεια σε γειτονικέ χώρες για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρήπανσης. Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με τι άλλο και εγώ τοποθετήθηκα πάρα πολύ επιφυλακτικά και αναφέρω μόνο επανειλημμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτέλους μια μελέτη σκοπιμότητας να δούμε που να ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Πριν γίνει αυτό δεν μπορεί κανείς υπεύθυνα να ψηφίσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Σας προτείνω λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει 25% δικαιώματα ψήφου, δηλαδή με τι άλλο δικαίωμα άρνηση κυρίας ή δυνατότητα σε ό,τι αφορά τις ε, νιοψίες, τις επιθεωρήσεις, αλλά και την επιλογή του διορισμού του εκάστοτε διευθυντή. Ολοκληρώνω με τις εξής παρατηρήσεις. Γνωρίζω ότι έχουμε διαφορές με το Συμβούλιο και θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς και αν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών μας έστειλε ένα μήνυμα ότι δεν είναι τόσο άκαμπτοι στη θέση τους, αλλά έχουν βάλει λίγο νερό στο κρασί τους. Αλλά και πάλι είναι συνέργειες αυτές. Θα πρέπει όμως αυτά που αποφασίσουμε να τα εφαρμόζουμε και στις χώρες μας. Επίσης, εάν κάπου προστίθεται μια δραστηριότητα, είτε συμβουλευτική, είτε άλλη, είτε αρμοδιότητα. Να μην το καταστρέφουμε από την αρχή επειδή δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη. Ε, άμα είναι καινούργια τα καθήκοντα πρέπει να τη βρούμε, να τη φτιάξουμε την πραγματογνωμοσύνη, αφού είναι κάτι νέο. Και για το χρονοδιάγραμμα το τελευταίο, 21 Ιουνίου, συγγνώμη σήμερα είναι, στις 29 είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και το Σεπτέμβριο θα έχουμε δεύτερη συνεδρίαση με τους σκιώδες ηγητές. Έχω προγραμματίσει και τρίτη και ε, στη συνέχεια θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Κραντές για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά για τη σημερινή σας εξήγηση και για τη στάση σας. Επανειλημμένα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας και σας ευχαριστώ. Και μπορεί να καταλήξει σε κάτι θετικό, σε μια συνέντευξη θετική για όλους με τη συνδρομή όλων. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της έκθεσης γιατί θα έχουμε χρόνο σε επιμέρους τροπολογίες να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα. Καταρχάς εγώ θέλω να κάνω μια αξιολόγηση θετική για τον οργανισμό, για την ασφάλεια στη θάλασσα ως οργανισμό. Νομίζω ότι με το χρόνο ο οργανισμός αυτός, με την πάροδο του χρόνου, ε, απέκτησε κάποιο κύρος. Γιατί είναι πολύ καλή διαχείρισή της. Η δράση της σημαίνει ε, εξοικονόμηση χρημάτων για τα κράτη-μέλη και προστιθέμενη αξία. Γιατί έχει κύρος, δεν είναι μόνο ένα γραφειοκρατικό εργαλείο που ανέκαθεν η Επιτροπή μας ε, αποστρεφόταν και απέριπτε. Ε, είναι πολύ καλή η διαχείρισή της και δεν θα πρέπει να αλλάξει. Και εδώ επικρατούν τρεις αρχές. Πρώτον, δρά κατόπιν ετήσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατών μελών. Δεύτερον, ουσιαστικά εκτελεί αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τρίτον δεν προσπαθεί να αποφύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Επιτροπής μας. Υπό την αυτή Πρόεδρε νομίζω ότι αυτές οι τρεις αρετές που σας ανέφερα δεν πρέπει να χαθούν. Θα ήταν κίνδυνος ο Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα να θελήσει να αυτονομηθεί ε, να ανεξαρτητοποιηθεί κατόπιν αυτής της επιτυχίας. Για μένα αυτό είναι κίνδυνος και απειλή. Λοιπόν, θα πρέπει να εξορπηθεί το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου υπερεκπροσωπούνται τα κρατημέλη βάρος της ευρωπαϊκή Επιτροπής, όπως είπε και ο εισηγητής. Δεύτερον, θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει αυτόνομη ε, εντολή για λήψη αποφάσεων, ε, εκτελεί αυτά που τις λένε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης υπάρχει μια σύγκρουση κομισιών κρατών μελών και θα πρέπει να λυθεί αυτό. Έχουν δίκιο τα κρατημέλη από το Τιμιά που λένε ότι επειδή ζούμε χαλεπούς καιρούς θέλουν να κάνουν οικονομίες και περικοπές και να αποφεύγουμε έξοδα που δεν έχουν προστιθέμενη αξία. Τα είπε και ο εισηγητής αυτά. Αλλά από την άλλη πιστεύω ειλικρινά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο. Ότι η διακυβέρνηση δεν μπορεί να χαθεί από τα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί θα ήταν αβέβαιο το αποτέλεσμα. Αξιολογούμε θετικά το έργο του εισηγητή και την έκθεση. Θα έχουμε χρόνο για τις τροπολογίες όπως σας είπα και με την επιφύλαξη ότι οι τροπολογίες θα είναι θετικές. Για κοινέ θέσει. Το Συμβούλιο μπορεί να έχει επιφυλάξει και δικαιολογημένε και θεμητέ, αλλά να τις συζητήσουμε για να μην οδηγηθεί σε παράλυση ο οργανισμός αυτός. Να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν περισσότερες εξουσίες και ε, να είναι αποτελεσματική η δράση για να μην ε, παραλύσει ή να μην επιβραδύνει την ευρωπαϊκή πορεία. Και σήμερα μπορεί να είναι απλουστευτικό αυτό που λέω, αλλά όταν κάποιο είναι ευρωπαϊστή, είναι υπέρ τη Ευρώπη, σημαίνει ότι είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αυτή θέλει να προωθεί την Ευρώπη. Ε, εγώ ήμουν εισηγητή στο ΕΡΙΚΑ, στον κανονισμό και στην οδηγία. Είναι παλιά υπόθεση αυτή. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριμένες ε, δράσεις αναθέσει στον οργανισμό. Να κάνει νιοψίες ο οργανισμός, αλλά δεν πρέπει να χάσει ε, την αρμοδιότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απέναντι στους νιογνώμονες, στις αναγνωρισμένους ε, οργανισμούς, οι οποίοι αγωνίζονται να ε, αναμειχθούν στο άρθρο 10 για την αμοιβαία αναγνώριση και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, η εφαρμογή του κανονισμού και η ε, παρακολούθηση θα πρέπει να είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το τεχνικό σκέλος και το πολιτικό ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για ε, τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ο κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 17. Διακυβέρνηση. Είναι Καλή η πρόταση του εισηγητή, μπορούμε να την δεχτούμε, να συμμετέχουν ε, ισορροπημένα τα τρία θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο για τον εκτελεστικό διευθυντή ε, και θα είναι επίσης αποδέκτη στο Κοινοβούλιο. Ε, σε ό,τι αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία, τα ποτάμια, μπορεί το θέμα αυτό να είναι πολύ προσφυλές αλλά νομίζω ότι είναι μια δημοσιονομική περιπέτεια για σήμερα. Το είδαμε και στην έκθεση Στέρξ. Λοιπόν, για τις εξέδρες εξόριξης καταλαβαίνετε ότι θα είναι επίμαχο. θα πρέπει να είμαστε τολμηροί. Μπορούμε να βρούμε νομική βάση και η ίδια η έκθεση του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου μιλάει για εγκαταστάσεις. Εγώ συμφωνώ με τη θέση του εισηγητή. Βεβαίω και το είπε και ο συγητή, όταν διευρύνεται η εντολή θα πρέπει να διατίθεται και μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και να πούμε στο Συμβούλιο ότι υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να βάζουμε και το χέρι στην τσέπη καμιά φορά γι' αυτά. Αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ τον εισηγητή και επιφυλάσσομαι να κάνω τροπολογίε ε, για να βοηθήσουμε να εξυπηρετήσουμε το γενικό στόχο της κοινή ε, πορείας και της συνένεσης που νομίζω ότι είναι εφικτός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλέκενστάιν για την έκθεσή του και να του πω ότι θα εργαστούμε από κοινού για να συμφωνήσουμε σε γενικές γραμμές. Συμφωνώ με τα όσα είπε και ο ίδιος και για να μην επαναλάβω θέματα που έχουμε πει σε άλλες επιτροπές, πρέπει να σας πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ε, μεταξύ άλλων για να είμαστε συνεπείς με αποφάσεις του Κοινοβουλίου μας ε, ο κύριος Γκράντες ε, Πασκουάλ μίλησε και για τη δική του έκθεση, αλλά έχουμε και την έκθεση του κυρίου Κόλ, την έκθεση του κυρίου Στέρξ, την έκθεση της κυρίας Μάισνερ για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και γενικότερα αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Ό,τι κάνουμε τώρα είναι ε, απόλυτη συνέχεια των όσων ε, κάναμε στο παρελθόν. Ό,τι κάνουμε στην έκθεση αυτή λοιπόν θα πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου, αλλά πραγματικού ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου. Γι' αυτό τι θα μας επιτρέψει, τα εξής δύο. Πρώτον, να είμαστε αποτελεσματικοί στη δράση μας, στην αντιμετώπιση της ε, θαλάσσιας ρήπασης από πλοία και χωρίς καμία αμφιβολία θα πρέπει επίσης να ε, προσθέσουμε εγκαταστάσεις εξόριξης ή διερεύνησης για πετρέλαιο φυσικό αέριο. Γιατί αν αύριο έχουμε πρόβλημα με μια εξέδρα εξόριξη πετρελαίου, τι θα κάνουμε δηλαδή. Επειδή δεν είναι καράβι. Τι, τι ε, εργαλεία έχουμε και μέσα. Ποιος θα το συντονίσει. Ποιον θα καλέσουν τα κράτη-μέλη. Ας μην περιμένουμε άλλη μια φορά να γνωρίσουμε τέτοια κρίση για να αρχίσουμε να το σκεπτόμαστε και να διευρύνουμε με αποφασιστικό τρόπο τις ε, αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ. Λοιπόν, να είναι ένας ευρωπαϊκός θαλάσσιος χώρος, να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε κρίσεις μπορούμε να έχουμε ανα πάσα στιγμή και δημιουργώντας αυτό το χώρο θα διευρύνουμε και την αποτελεσματικότητα και την υπηρεσία και προς τίτες χώρες, γειτονικέ χώρες. Και ε, συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέει ο συγητής. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο εντός αυτού του χώρου και της αποτελεσματικότητας να δημιουργήσουμε ένα ε, δίκτυο ε, σχολών ναυτικών για την εκπαίδευση κάποιο κράτος ε, και κάποιες οργανώσεις με τρόμαξαν γιατί είπαν ότι η έννοια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας ταυτίζεται με μια ενιαία ευρωπαϊκή έδρα. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Δεν είπαμε να γίνει κάπου μια σχολή ναυτικών και πουθενά άλλου. Ένα δίκτυο για να είναι εναρμονισμένη εκπαίδευση, κατάρτιση των ναυτικών στα κράτη-μέλη για να μπορούμε να δρούμε και πιο αποτελεσματικά. Γιατί Όλες οι χώρες μπορεί να πληγούν. Επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκό ε, ενιαίο θαλάσσιο χώρο, ε, διεύρυνση της εντολής να καλύπτει και τις εξέδρες εξόριξης, εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών και για την ευρωπαϊκή εκτοφυλακή. Συμφωνώ. Συμφωνώ και με αυτά που είπε ε, ο εισηγητής. Περιμένουμε την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποφασίσουμε οριστικά. Ξέρουμε ότι έχουμε κρίση, αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά να ακούμε τέτοια δημοσιονομικά επιχειρήματα που μας το κοπανάνε συνέχεια και το Συμβούλιο και οι πάντες για να αποφύγουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία για περισσότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Εμεί θα πρέπει να προχωρήσουμε, θέλουμε πραγματικά. Να δώσουμε ευρωπαϊκές απαντήσεις. Και στο θέμα της διακυβέρνησης θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ισορροπημένη στάση, όπως προσθέτει και ο, ο πρόεδρος, ο εισηγητής, συγγνώμη. Χάθηκε αυτό τελευταία. Δεν συμφωνώ με το Συμβούλιο που θέλει να ε, έχει μισιακή σχέση ή προνομιούχα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς θα κάνουμε και τροπολογίες ως ομάδα προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ πρόεδρε όχι μόνο οι παρόντες εδώ, αλλά και οι πιστή φίλοι μας από το webstream γνωρίζει ότι η ομάδα μου ε, είναι επικριτική απέναντι στους διάφορους οργανισμούς με διάφορες αρμοδιότητες, καθήκοντα και χρήματα που πάνε στους οργανισμούς αυτούς. Αυτό συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να σας πω ότι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα βεβαίως μπορεί να έχει κάνει κάποια θετικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Το ε, είδαμε. Και τι σημαίνει αυτό για τη θάλασσα και για την αυσιπλοεία. Αλλά τι βλέπουμε με την παρούσα πρόταση και με τις τροπολογίες. Ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή τώρα. Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΜΣΑ ως θεματοφύλακας ή ως χωροφύλακας. δηλαδή, ε, το να κάνει τώρα επιθεωρήσεις δεν ξέρω αν συνάδει με ε, το ρόλο του ΕΜΣΑ ή τι έχει να κάνει με τη πιστοποίηση και με την κατάρτιση των ναυτικών. Τι δουλειά έχει η ΕΜΣΑ εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά ε, τον κλάδο ε, των ε, ναυτικών, των εργαζομένων, των πλειοκτητών, των ιογνωμόνων, αλλά όχι για την ΕΜΣΑ. Και επίσης η ακτοφυλακή. Είναι σαν να βγάζεις κόκκινη κάρτα στα λιμενικά σώματα και στην ακτοφυλακή που υπάρχει σήμερα. Ε, σαν να τους λες ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας και σας τραβάμε τα αυτή. Εγώ δεν έχω καμία ένδειξη ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και υπάρχει το μνημόνιο, λέει, του Παρισιού. Ε, αυτό είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία που κάνει λιμενικούς ελέγχους και πάρα πολύ καλά. Γιατί να το καταργήσουμε και να το δώσουμε στην ΕΜΣΑ. και για την εσωτερική ναυσιπλοεία θα ήθελα να μας ενημερώσει ή να μας διαφωτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει να κάνει νιοψίες και επιθεωρήσει η ΕΜΣΑ και ούτε στην εσωτερική ναυσιπλοεία, διότι αυτό είναι ε, εθνική υπόθεση. Και οι νεογνώμονες μπορούν να ταξινομούν και να αξιολογούν και ε, τα ποταμόπλια. Ε, όχι μόνο τα πλοία που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Και δεν μην ανακατεύεται η έμσα εκεί. Αυτά ήθελα να ακούσω λίγο από τον κύριο Καραμίτσο. Και επιστρέφω στην αρχική μου τοποθέτηση. Πολύ επικριτικά και ε, ε, επιφυλακτικά βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν και ανάλογα θα καθορίσουμε και τη στάση μας στην ψηφοφόρια. Ευχαριστώ. Κύριο Στέιλορ. Thanks, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν γέννη συμφωνούμε με την έκθεση και την προσέγγιση του κ. Φλέκενστάιν. Θεωρούμε πως είναι θετική και περιστατωμένη. Είναι επίκαιρη η στιγμή να αναθεωρηθεί ο ρόλος της ΕΜΣΑ με πιθανή ε, επέκταση της εντολής της, αλλά Πιστεύω ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν επικαλύπτουμε οποιασδήποτε ευθύνε, ανάμεσα στην ΕΜΣΑ δηλαδή και άλλες ε, υπηρεσίες, άλλους οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως θα υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι ώστε η ΕΜΣΑ να μπορεί να εκτελέσει τις ε, αρμοδιότητές της. Συμφωνούμε ότι με την προσέγγιση της Κομισιόν ότι θα πρέπει δηλαδή να εξετάσουμε τις δυνατότητες ε, κάλυψης. πριν να εισάγουμε οποιαδήποτε πολιτική. Νομίζουμε πως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του θαλασσίου και παρακτήου περιβάλλοντος και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι τα τμήματα της έκθεσης που ασχολούνται με το πετρέλαιο και τις ε, πλατφόρμες εξόρυξης στην ανοιχτή θάλασσα χρειάζεται να ενισχυθούν. Επίσης και ο στόλος επίγουσας ανάγκης για να έχει πρόσβαση ε, για διάσωση πλοίων για την πρόληψη της μόλυνσης και εκεί χρειάζεται ενίσχυση των παραγράφων. Θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες στην έκθεση αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για την έκθεσή του, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές. Είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, πόσο μάλλον που ε, οι ναυτιλιακές μεταφορές ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο, τα τελευταία δέκα χρόνια θα αυξηθούν κατά 20%. Και θα πρέπει να έχουμε κατά νου μας ε, τις διαφορετικές ε, χρήσεις της ε, θάλασσας γύρω μας. Για παράδειγμα, εάν έχουμε ένα μεγάλο, κάποια μεγάλη ζημιά, είτε είναι σε κάποιον ανεμόμυλο, είτε σε εξαδρεξόξης πετρελαίου και είτε αυτό γίνει στη Βόρεια Θάλασσα ή στην Μεσόγειο. Θα πρέπει η, μονάδες ε, επίγουσας παρέμβασης ε, να συντονίζονται μεταξύ του Η ΕΜΣΑ εποπτεύει αλλά θα πρέπει ε, τα σκάφη να έχουν τις τεχνικές προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό το κάνουμε με εθνικούς φορείς κλπ. Θα πρέπει όμως να γίνει και αυτός ο συντονισμός και γι' αυτό η ερώτησή μου είναι στρατηγικά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Μιλάμε για τα επόμενα 10 χρόνια, μιλάμε πάντα για τη στρατηγική 2020. Ε, αυτή η στρατηγική δεν συνδέεται μόνο με την ε, ε, ε μείωση των εκπομπών και με ε, περιβαλλοντικά θέματα, έχει να κάνει και γενικά με το θέμα των ε, ασφαλών μεταφορών στη θάλασσα. Στο Βόσπορο ή στη Βαλτική υπάρχουν ε, διάφορες κρίσιμες καταστάσεις ε, με τα ραντάρ. Έχουμε συζητήσει και τα διάφορα συστήματα με δορυφορική ε, βοήθεια, με, βάση το Γαλιλαίο, πόσο καλά είμαστε εξοπλισμένοι. Ο τουρισμός στις ακτές μας παίζει επίσης ρόλο. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε ε, σημαντικά ατυχήματα. Θα πρέπει να εργαστούμε προληπτικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Προτού να δώσω το λόγο στην κυρία Μάισνερ, να καλωσορίσουμε μια ομάδα προσκεκλημένων ε, της κυρίας Μάισνερ. Έχουν, ε, έχουν καταφτάσει από την κάτω Σαξονία. Ε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είναι ομάδα κατάρτισης ενηλίκων. Ε, ελπίζω να ε, ε, ευχαριστηθείτε την επίσκεψη ε, της... Ε, έχετε το λόγο κύριε Μάστερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα καν δει ότι κατέφτασε η ομάδα αυτή. τρία θέματα θα ήθελα να θίξω. Το πρώτο είναι η ρήπανση των θαλασσών που μπορεί να ελεγχθεί όχι μόνο από τα ε, πλοία αλλά και από πλατφόρμες. Θα πρέπει να προσέξουμε τα οικοσυστήματα και ήδη πέρσι στην ε, σχετική μου έκθεση ανέφερα ότι τα οικοσυστήματα αυτά θα πρέπει να προστατευτούν. Ε, στην ε, γη έχουμε 70% θάλασσα και 30% γη. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε στη θάλασσα να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε στη γη. Στην ξηρά. Ε, επίσης, ε, όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Φαντάλεν, ε, από ό,τι κατάλαβα, ο εισηγητής δεν θέλει να αναλυφθεί η εκπαίδευση από την ΕΜΖΑ, αλλά να γίνει η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Η ΕΜΖΑ σίγουρα έχει ιδέες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κατάρτιση των ναυτικών. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Και η τελευταία μου παρατήρηση αφορά την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Εδώ και πολύ καιρό εδώ ζητάμε εδώ στο Κοινοβούλιο μελέτη ε, σκοπιμότητας. Η Κομισιόν δεν έχει κάνει τίποτα. Ε, και στην ε, έκθεσή μου θύμισα ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. πρέπει κάτι να γίνει και γι' αυτό βρίσκω χρήσιμο ότι ο κύριος Φλέγκενσταν έχει συμπεριλάβει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Mm. Ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να στηρίξω κάποια από τα όσα ανέφερε ο συνάδελφος Πίτερ Φαντάλεν όσον αφορά τον οργανισμό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, θετικές, πολλά θετικά στοιχεία στη δημιουργία της υπηρεσίας, ε, πρότυπα ασφαλείας στην εργασία, διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες σαφώς είναι πολύ θετικές και νομίζω πως είναι λογικό να βάλουμε εκεί όπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει επικάλυψη. Ε, επίσης, όσον αφορά τη δική μου αντιπροσωπεία, όπως σας είπα, εν γέννη είμαστε θετικοί και χωρίς να χρειάζεται να μπω τώρα σε όλες τις τροπολογίες που είναι αρκετές, υποστηρίζουμε την 5 για το, την παράκτια ναυσιπλοεία είναι πολύ ε, θετικό. Μια τροπολογία επίση είναι η τροπολογία 3 που αφορά την αύξηση του προπολογισμού, αλλά νομίζω πως αυτή την περίοδο τεράστιων περιορισμών η ΕΜΣΑ είδε σημαντικές αυξήσει, σημαντικές ε, θέσεις απασχόλησης και νομίζουμε ότι τα χρήματα τώρα πρέπει να ιεραρχηθούν και να πάνε σε κάποιου άλλου τομείς στον προπολογισμό τη Κομισιόν. Δεν είμαστε σε θέση λοιπόν να αρχίσουμε να ψάχνουμε χρήματα, μάλλον νέα φρέσκα χρήματα βασικά. Θα πρέπει πολύ σοβαρά να το σκεφτούμε από πού θα έρθουν ε, έξτρα χρήματα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ε, το θέμα των παρακτήων, ε, των, ε, της ακτοφυλακής, με συγχωρείτε, Υπάρχουν ρυθμίσεις, για το Frontex, ε, για, για, για τις ε, διάφορες ακτοφυλακές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως γιατί πολλοί, πολλές, ε, πολλά καθήκοντα έχουν οι ακτοφυλακές τη σήμερα ημέρα, όχι μόνο πολιτικά αλλά και στρατιωτικά και δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα καθόλου. Περαιτέρω λοιπόν συνεργασία θα πρέπει να υπάρξει όντω για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τελευταία μου παρατήρηση αφορά τον ρόλο της ΕΜΣΑ για τη διερεύνηση των ατυχημάτων. Τροπολογία 17, νομίζω πως η Κομισιόν έχει δίκιο εδώ ε, σε σχέση με την αρχική παρατήρηση. Η θέση αυτή θεωρούμε πως είναι σωστή γιατί ειλικρινά δεν πιστεύω πως ο οργανισμός έχει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την αντιμετώπιση ατυχημάτων και την διερεύνηση αυτών. Εν γέννη, Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, έκανε πολύ σκληρή δουλειά. Απλώς θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση σε κάποιους τομείς. Για γέννη υπάρχει συνένεση για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Η ρήπανση είναι κάτι που μας αφορά όλους σοβαρά. Έχουμε πολύ καλή βιομηχανία πετρελαίου στα ευρωπαϊκά ύδατα. Ε, είναι λοιπόν αφορά την καλύτερη συνεργασία και την ε, μη επικάλυψη. Ο κ. Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον ε, μελετάμε το υποσυζήτηση κείμενο για τον οργανισμό της ΕΜΣΑ. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Η ΕΜΣΑ έχει κάνει θετικό έργο και αναφυσβήτητα προσδίδει προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια της Ένωσης να εφαρμόσει την ε, πολιτική των θαλασσίων μεταφορών. Και βεβαίως έχει έναν όχι αμεληταίο συντονιστικό ρόλο. Αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να επιδιώξουμε στο κείμενο αυτό είναι η περαιτέρω ποιοτική βελτίωση και ευάθυνση των ήδη υπαρχουσών αρμοδιοτήτων που έχει. Να τις κάνουμε καλύτερες, να τις εμβαθύνουμε περισσότερο. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και των αποστολών της είναι ένα άλλο ζήτημα. Και πάντως, όταν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, διότι είναι προφανές ότι δεν πρέπει να κάνουμε την έμσα, δεν πρέπει να την αφήσουμε να μετατραπεί σταδιακά σιγά σιγά σε ένα sui generis νιογνώμονα ή σε ένα sui generis εκπαιδευτικό κέντρο ναυτικών είτε σε μια sui generis ακτοφυλακή. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πώς αυτά τα βήματα θα γίνουν ώστε να μην δημιουργήσουμε μια νέα περίεργη ε, θεσμική μορφή αλλά να μείνουμε σταθερά στις αρμοδιότητες που αυτός ο οργανισμός έχει να επιδιώξουμε να τις κάνουμε καλύτερες και αποδοτικότερες για να συνεχίσει να παράγει αποτελεσματικά και να δίνει την προστιθέμενη αξία που αναφυσβήτητα έχει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι μια γενική παρατήρηση. Θα εξειδικευθεί και με τις συγκεκριμένες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. For the commission, Mr. Ευχαριστώ. Από την Κομισιόν ο κύριος Καραμίτσος. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή καθώς και ολόκληρη την Επιτροπή σας που βασικά μας έκανε θετικά σχόλια για την έμσα. Είμαστε πολύ ευτυχείς με την δουλειά που έχει γίνει για τα κρατη και για την Επιτροπή για την εποπτεία και την επαλήθευση όλης της νομοθεσίας αυτής. Πιστεύω λοιπόν πως ε, από αυτή την άποψη εγώ θα έπρεπε να συμφωνήσω με τον τελευταίο μιλητή ότι δηλαδή θα πρέπει να δούμε πόσο περισσότερο μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της απόδοσης, την εμβάθυνση αυτής της δουλειάς αλλά και να δούμε τι επιπλέον καθήκοντα τι μπορούμε να θέσουμε στην ε, υπηρεσία αυτή, στον οργανισμό αυτό. Και σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή αλλά και τα άλλα μέλη που είδαν τα ωφέλη αυτής της πρότασης. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε στο maximum δυνατό την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε ώστε να μας βοηθήσουν εκεί με προστιθέμενη αξία ε, για καθήκοντα, για πράγματα που θα πρέπει να γίνουν από την άποψη της ναυσιπλοείας. Από αυτήν την άποψη λοιπόν η επέκταση των καθηκόντων θα πρέπει να σχεδιαστεί με πολύ προσεκτικό τρόπο και προσπαθήσαμε αυτό να το κάνουμε ώστε να έχουμε το maximum όφελος από την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε. Από αυτήν την άποψη λοιπόν η πτυχή της, του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, της συμβατότητας ανάμεσα στα συστήματα ναυσιπλοείας, ε, στις πλωτές οδούς και στην ε, θάλασσα, η, η, η συντονισμός των νεογνωμόνων κτλ. Όλα αυτά είναι δραστηριότητες που κάνουμε χρησιμοποιώντας το προσωπικό και την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε. Και από αυτή την άποψη τα περισσότερα θα βασιστούν στην αναδίπλωση των εσωτερικών πόρων και κάποιου επιπλέον πόρου, κάτι πολύ περιορισμένο. Δηλαδή, μιλάμε για 5% αύξηση των πόρων για τα επιπλέον αυτά καθήκοντα. Δεν είναι τίποτα σημαντικό αν συγκρίνει κανεί τα ωφέλη. Ε, Έχουμε ένα δύο θέματα. Το ένα είναι η διαχείριση και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε την ισορροπία. Να σας θυμίσω μόνο απλά ότι στο αρχικό κείμενο που υιοθετήθηκε τότε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν τη διεύρυνση, προέβλεπε τουλάχιστον 20% παρουσία των εκπροσώπων της ε, ε, Κομισιόν. Από την άλλη πλευρά, ε, θα πρέπει να μείνουμε στο πλαίσιο της ασφάλειας, γιατί πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Ναυσιπλοίας και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά τις ε, πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και την ανοιχτή θάλασσα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν κάτι συμβεί, αν γίνει κάποιο τύχημα, υπάρξει ρήπανση και σήμερα οι περισσότερες πλατφόρμες ε, βρίσκονται στη βόρεια θάλασσα, στα βόρεια της Ευρώπης δηλαδή. Από την άλλη πλευρά έχουμε πολλά πλοία κατά της ρήπανσης που βρίσκονται στο νότο. Ε, θα πρέπει να δούμε δηλαδή πώς... Ε, θα κατανείμουμε αυτούς τους πόρους ώστε να μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία για αυτές τις περιπτώσεις. Να καλύψουμε δηλαδή όχι μόνο ρήπανση από την αναψυπλοή αλλά και από τις εξέδρες πλατφόρμες εξόριξης. Τώρα, να πάμε να προσθέσουμε όλα αυτά ε, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί δεν έχουμε πρωτογενή νομοθεσία. Αυτό που κάνουμε με τις ε, εταιρείε αυσιπλοείας και αυτό που κάνουμε με τα κράτη-μέλη, τους γνώμονες αλλά και ε, τα εκπαιδευτικά Ινστιτούτα σε ολόκληρο τον κόσμο, τους στέλνουμε εκεί και ξέρουμε, έχουμε μια πρωτογενή νομοθεσία και ξέρουμε τι θα επιθεωρήσουν. Από αυτή την άποψη όμως δεν έχουμε άμεση δικαιοδοσία να πάμε και να πούμε ναι θα πρέπει να πάμε να ελέγξουμε το τάδε μέρος. Από την άλλη πλευρά, άλλοι τόνισαν ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμό ανάμεσα στους οργανισμούς. Και ως προς αυτό μιλάμε για θαλάσσια ρήπανση. Εμείς από την πλευρά μας λέμε ότι η ναυσιπλοεία δημιουργεί, προκαλεί θαλάσσια ρήπανση. Η έμσα θα πρέπει να εξετάζει και την ρήπανση στην ξηρά που προκαλείται από τις θάλασσες. Δεν το έχουμε ακόμα αυτό τη δυνατότητα. Μην επεκτείνουμε δηλαδή το ρόλο της ΕΜΣΑ πέρα από την αυσιπλοεία. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Και μετά υπάρχουν και ένα-δυο άλλα πράγματα, όπως το, το θέμα της ακτοφυλακής. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ήδη σήμερα η ΕΜΣΑ έχει θεσπίσει ήδη δοδούς συνεργασίες. Για το τρίτο πακέτο ναυσιπλοείας, ας πούμε, για την παρακολούθηση των σκαφών, το δίκτυο ασφαλείας, το... Ο εντοπισμός και ανείχνευση σε μεγάλη εμφέλεια. Όλα αυτά ήδη τα έχουμε κάνει και έχουμε διευκολύνει το συντονισμό των πόρων των κρατών μελών. Περισσότερα μπορούν να γίνουν και ναι, σας χρωστάμε μια έκθεση, είναι αλήθεια. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την μελέτη, αλλά δεν είχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα και ξεκινήσαμε άλλη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. για τις επιθεωρήσεις. Νομίζω πως είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός των ρόλων ανάμεσα στην ε, επιθεώρηση και την αξιολόγηση. Η ΕΜΣΑ είναι το σώμα που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη και κομισιόν για να επιθεωρούν τα συστήματα των συνεχνόμενων τρίτων χωρών. Αλλά η ίδια η αξιολόγηση και η τελική επαλήθευση του τι συμβαίνει ε, γίνεται. Δεν γίνεται από εμά. Αυτό του είδου ο διαχωρισμό θα πρέπει να διατηρηθεί και ο εισηγητή συμφωνεί με αυτό νομίζω. Πιστεύουμε, λόγω της σύγκλησης απόψεων της Επιτροπής αυτής και το γεγονός ότι έχουμε απομακρυνθεί από την αρχική αρνητική άποψη του Συμβουλίου, δεν νομίζω πως απέχουμε και πολύ από την τελική συμφωνία με μια πρώτη ανάγνωση, με λίγη καλή θέληση από το Συμβούλιο, ώστε να διορθωθούν κάποιες από τις τα τελευταία λαθάκια που ξέφυγαν, όπως για παράδειγμα το γεγονός πως ήδη στο αρχικό κείμενο τα κάτι μέλη είχαν την υποχρέωση να βοηθούν ε, την ε, οργανισμό όταν ο οργανισμός θα τους επιθεωρούσε, θα τους ε, έλεγχε. Αυτό έχει εξαφανιστεί από το κείμενο χωρίς λόγο με πάση περιπτώσει, τα κράτη-μέλη δουλεύουν, ε, συνεργάζονται με τον οργανισμό εδώ και χρόνια και στηρίζουν τους επιθεωρητές. Γιατί να το αφαιρέσουμε λοιπόν. Έπειτα υπάρχει το ζήτημα της έρευνας και ανάπτυξης και εδώ χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τον οργανισμό όχι ως ε, διευθυντή έρευνας, αλλά τουλάχιστον να είμαστε σε θέση να ορίσουμε τι χρειαζόμαστε να κάνουμε πώς αυτό θα ενταχθεί στην πτυχή των ορισμών της νομοθεσίας στη συνέχεια. Είναι ένας βοηθητικός ρόλος προς τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Αυτά τα δύο θέματα λοιπόν είναι δύο παραδείγματα που εξεφανίστησαν από το κείμενο και μπορούμε να τα ξαναβάλουμε χωρίς δυσκολίες. Έπειτα, για την επέκταση των Αρμοδιατήτων της, ε, του οργανισμού υπήρχαν διάφορες ρήτες ασφαλείας ε, και θα ήταν υπερβολικά γραφειοκρατικό και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας προς όφελος της βελτίωσης της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Εγώ προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδης ώστε να βελτιώσουμε το κείμενο και ελπίζω ότι μετά από την ψηφοφορία τον Οκτώβριο θα καθίσουμε μαζί με την Προεδρία για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για να βρούμε μια συμφωνία στην ε, πρώτη ανάγνωση, γιατί ξέρουμε και ότι η Πολωνική Προεδρία θέλει να προχωρήσει το θέμα. Ευχαριστώ και θα περιμένουμε τις ε, τροπολογίες και θα συνεργαστούμε μαζί σας ώστε να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως λέω πάντα, είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με τις προεδρίες και εάν οι προεδρίες ήταν λίγο πιο δεκτικές απέναντι στις θέσεις ε, του Κοινοβουλίου ε, σε κάποιες περιπτώσεις ε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Πάντα με εκπλήσει που οι προεδρίες λένε ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα και να ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας και κατόπιν ε, διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα που συναντούμε προέρχονται από το Συμβούλιο Υπουργών. Ε, θα το έχουμε όμως κατά νου. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φλέκενστάιν αν έχει κάτι να προσθέσει. Ναι κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Κύριε Φαντάλεν, συγγνώμη, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο πολύ σωστά είπατε. Φυσικά ήδη υπάρχουν ε, έλεγχοι στα λιμάνια. Το ερώτημα είναι, μπορούμε με καλύτερο συντονισμό μέσω της ΕΜΖΑ, μπορούμε σε συνεργασία με την ΕΜΖΑ να λύσουμε πιο αποτελεσματικά το θέμα και μπορούμε να ε, πετύχουμε αποτελέσματα από τη συνέργεια στα διάφορα κράτη-μέλη. Και μόνο αν η απάντηση είναι ναι, τότε έχουν όλα αυτά νόημα. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. η επικάλυψη εργασιών δεν ενδιαφέρει ούτε εμένα. Δεύτερον, σας παρακαλώ να εξετάσετε λίγο πιο προσεκτικά την διαφορά ανάμεσα στις δραστηριότητες και τις συμβουλευτικές εργασίες. Η ΕΜΖΑ δεν θα έχει δικά τις δικές της σχολές. Νομίζω όμως ότι μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τα ε, τα κράτη-μέλη και την ε, Κομισιόν μέσω των συμβουλών της. Τρίτο θέμα. Όσον αφορά το πρόγραμμα Blue Belt, το θέμα εδώ δεν είναι να επιβάλλουμε ε, ένα καθήκον στην ΕΜΣΑ. Το ίδιο το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2010 αποφάσισε ότι χρήσιμο είναι στο πρόγραμμα Blue Belt να συμμετάσχει και η ΕΜΖΑ στην εκπόνηση. Σίγουρα κάποια στιγμή θα προκύψει το ερώτημα αν όλα αυτά στοιχίζουν ε, περισσότερα χρήματα. Αυτό εξαρτάται από το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που ε, προτείνουμε εδώ. Και το αν ε, εκμεταλλευτούμε τις πιθανότητες συνέργειας που υπάρχουν. Στις προτάσεις που έχουμε εδώ μπροστά μας δεν βλέπω καμιά υπερβολική διεύρυνση των καθηκόντων της ΕΜΖΑ. Ε, το πολύ πολύ να μιλάμε για προσεκτικές ε, διευρύνσεις, προσπάθειες διεύρυνσης, αλλά θα παρακαλούσα να δούμε, ε, να έχουμε κατά νου την συνολική προοπτική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι χρήσιμο μαζί στο θέμα αυτό. Ε, και νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολε οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Το, Συμβούλιο, η Πολωνική Προεδρία, ε, νομίζω ότι... Ε, νομίζω ότι μπορούμε να του έχουμε εμπιστοσύνη και ότι θα πετύχουμε αυτά που προτείνουμε εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλέκενστάιν. Να θυμίσω στους βουλευτές ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 29η Ιουνίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Οκτώβριο και προβλεπόμενη ημερομηνία στην Ολομέλεια είναι ο Νοέμβριος. Αυτό λοιπόν είναι το χρονοδιάγραμμα. Ε, προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών 29 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Έτσι έχουμε ολοκληρώσει την εμείς διάταξη για σήμερα το πρωί και θα σας δω όλους στις 3 η ώρα για να συζητήσουμε τη Λευκή Βίβλο. Ευχαριστώ.